Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα πρέπει να αρχίσουμε. Καθίστε παρακαλώ στές σας. Να ξεκινήσουμε. Την έκτακτη αυτή παράταση της συνεδρίασης της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ που έλαβε χώρα χθες. Σας υπενθυμίζω, έκτακτη παράταση είναι αυτή της συνεδρίασής μας. Για να εξετάσουμε τις δημοκρατικές ε, διαδικασίες στην κεντρική Μεσόγειο και την επίπτωση των ε, κυμάτων προσφύγων. Θα ακούσουμε την άποψη της Ουγγρικής Προεδρίας που θα εκπροσωπείται εδώ από την αυτοεξοχότητα Πίτερ Γκέρκας, ε, μόνιμο αντιπρόσωπο της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Επίτροπο Μάλστρα. Την οποία καλοξορίζουμε στις εργασίες της Επιτροπής μας, τον Γενικό Γραμματέα Δημό, που είναι ο Γενικός Γραμματέας της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και επίσης έχουμε τον κύριο Ήλκα Λάτινεν, τον γνωρίζετε, εκτελεστικό διευθυντή της Frontex. Θα συζητήσουμε τα γεγονότα που όλοι παρακολουθούμε στενά, καθημερινά, στην Ιρυσία, στην Αίγυπτο και στη Λιβύη. Μια πρώτη ζήτηση έλαβε χώρα στο Στρασβούργο, στην περασμένη σύνοδο, και τώρα θα ενημερωθούμε για τα πιο πρόσφατα γεγονότα από την Προεδρία του Συμβουλίου, την Επίτροπη Μάρσον, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τον Διευθυντή της Λαϊτινέν. Επιμένω. Έχουμε μια έκτακτη παράταση της συνεδρίασης της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για μια μισή ώρα. Και γι' αυτό τονίζω τη σημασία του χρόνου που θα χρησιμοποιήσουμε. Συνήθως ξεπερνάμε το χρόνο μας. Επιμένω λοιπόν ότι θα πρέπει να προσέξουμε και να μπορέσουμε σε μια μισή να ολοκληρώσουμε την συζήτηση αυτή. I suggest that we are to hear from our Λοιπόν, προτείνω να ακούσουμε κάθε ένα από τους επισκέπτες μας πέντε λεπτά. Θα έχετε ένα πρώτο γύρο των συντονιστών ας πούμε δυόμιση λεπτά ο κάθε συντονιστής και μετά θα ανοίξουμε την συζήτηση για όλους τους βουλευτές που θέλουν να μιλήσουν. Θα προτείνω λοιπόν να ακούσουμε πρώτα την Ουγγρική Προεδρία που εκπροσωπεί ο πρέσβης Πίτερ Γιώργος, που εκπρόσωπο της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Προεδρία εκτιμά πάρα πολύ την ε, δυνατότητα αυτή να σας δώσουμε μια παρουσίαση για το τόσο πολύπλοκο και ευρύ θέμα και επίσης να ε, πούμε πώς συνεργάζονται τα θεσμικά όργανα. Δύο στοιχεία. Κάτι τυπικό. Ο πρόεδρος της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής έχει επίσης τον ίδιο χρόνο να μιλήσει όπως και ο πρόεδρος της ο εκπρόσωπος μάλλον της Προεδρίας. Συναντηθήκαμε όλοι πριν από πέντε μέρες. Η Ουγγρική Προεδρία οργάνωσε ένα επίσημο γεύμα όπου η Επίτροπος Μάρστον, ο Γενικός, Ευθυντής, Γενικός ε, Γραμματέας Δήμων και ο εκπρόσωπος Λαϊ της Frontex ήταν παρόντες για να συζητήσουμε την κατάσταση στην Βόρεια Αφρική. Θα αναφερθώ σε πέντε σημεία τα οποία η Προεδρία θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. μπορούσαμε μέχρι στιγμή ε, να δούμε ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούσε να αντιδράσει αν χρειαστεί με όλα τα θεσμικά όργανα. Είμαι σίγουρο όμω ότι ε, ο κάθε ένα από του συναδέλφου εδώ θα παρουσιάσει τι δικέ του απόψει. Είναι πολύ πολύπλοκη η κατάσταση και αν μιλήσουμε την προετοιμασία του επερχόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου που το θέμα είναι στην Διάταξη, θα πρέπει να δώσουμε δύο απαντήσεις. Η μία για την οικονομική κατάσταση και η άλλη για την κατάσταση στην Βόρειο Αφρική. Μέχρι στιγμή η Προεδρία αντέδρασε σε πέντε τομείς. Καταρχήν, οι επιπτώσεις της ε, εισόδου των προσφύγων από την Τινησία, στην Τινησία συγγνώμη, και ζητήσαμε από τη Μάλτα και την Ιταλία σε αυτό το δείγμα που σας είπα να μας πούνε πώς ήταν η κατάσταση. Το συμπέρασμα ήταν ότι προς το παρόν η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα απάντησαν κατάλληλα. Κινητοποιήθηκαν όλα τα αρμόδια όργανα και οργανισμοί. Η κατάσταση βρίσκεται λοιπόν υπό έλεγχο και η Κομισιόν και η Frontex θα σας πει παραδείγματος χάρη περισσότερες λεπτομέρειες. Το δεύτερο στοιχείο είναι βέβαια οι Ευρωπαίοι πολίτες πρόσφυγες. Στην Τρίπολη δεν έχουμε την προσωπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε έχουμε μια ηγετική χώρα με πρεσβεία εκεί. Η Ουγγρική Προεδρία δηλαδή προσπάθησε και νομίζω ότι λόγω του περιορισμένου δυναμικού με δύο διπλωμάτες που είχαμε εκεί, καταφέραμε, λέω, να εισαγάγουμε σωστούς ε, μηχανισμούς συντονισμού, ούτως ώστε να είναι ενήμεροι εκπρόσωποι των κρατών μελών και πάνω από το 80% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη μπόρεσαν να ε, ε, μεταφερθούν από τη Λιβύη και βέβαια η Ουγγρική Προεδρία δεν βοήθησε μόνο τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλων χωρών. Της Ευρώπης ιδίω. Η διπλωματική προστασία ε, δίνεται αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι οι αρχές της Λιβύης βρίσκονται σε επαφή μόνο με την Ουγγρική Πρεσβεία για τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στάση της πάτου εκπροσώπου κινητοποίησε και το κέντρο ενημέρωσης που αυτή τη στιγμή σε μόνιμη βάση ανταλλάσσει ε, πληροφορίες και αν χρειαστεί κινητοποιεί δυνατότητες μεταφορών για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να φύγουν από την Λιβύη. Χθες είχαμε δύο κύρια γεγονότα όσον αφορά την δράση και την αντίδραση. Καταρχήν επιτυχημένη δραστηριότητα του Συμβουλίου, ένα fast track για να επιβάλλουν οι κοινοτικέ επικυρώσεις στη Λιβύη και εκπρόσωποι κρατών μελών που είναι και μέλη στο Συμβούλιο Ασφαλείας δήλωσαν ότι αυτή είναι η πιο ταχεία αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επιβλήθησαν λοιπόν οι κυρώσεις, ισχύουν αυτή τη στιγμή η απόφαση του Συμβουλίου και ο σχετικός κανονισμός ισχύει ήδη και προς το παρόν φαίνεται ότι αυτή ήταν η σωστή αντίδραση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν χρειαστεί όμως, η Προεδρία είναι έτοιμη να ε, ξανααντιδράσει, αν χρειάζεται να διαβριθεί ο κατάλογος των καιρώσεων, να μειωθεί ή οτιδήποτε. Και επίσης, ε, όχι μόνο για λόγους άμεσης ασφάλειας αλλά και οικονομικούς λόγους έχουμε την επίπτωση της κρίσης στην τροφοδότηση με ενέργεια της Ευρώπης. Το Συμβούλιο Ενέργειας χθες ε, δημιούργησε μια ευρεία εικόνα της κατάστασης όσον αφορά τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου και η κατάσταση αυτή τη στιγμή δείχνει ότι η Ευρώπη έχει αρκετά αποθέματα και δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να υπάρχουν οποιαδήποτε έκτακτα μέτρα αλλά θα παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρέσβη, κύριε Γιώργο. Σας ευχαριστώ για τις προσπάθειές σας να είσαστε και σύντομος. Είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα κάνει και η Επίτροπος Μάρτσο που της δίνω το λόγο. Very Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε για αυτά τα ενθαρρυντικά λόγια. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ και φαίνεται ότι όταν χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα μπορούν να συνεργαστούν ε, όπως πρέπει, όπως ανέφερε και ο πρέσβης και μαζί με την Επιτροπή ΑΦΕΤ ενημερωθεί από τον Επίτροπο Φιούλε. Φαίνεται λοιπόν ότι σε αυτές τις έκτακτες περιστάσεις μπορούμε να συνεργαστούμε σωστά και με σπουδή. Ζούμε εξαιρετικά γεγονότα. Πρόκειται για μία φωνή, ομαδική φωνή για την ελευθερία εκεί όπου υπήρχε μεγάλο δημοκρατικό έλλειμμα, αλλά η κατάσταση στη Λιβύη μας απασχολεί και μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση ε, βράχη, μέσο και μακροπρόθεσμα και να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους αυτούς στην οδό προς τη δημοκρατία και να χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατό μέσο προς την επίτευξη αυτού. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπε ο πρέσβης ε, έγινε μία ιδιαίτερα καρποφόρα και επικοδομητική συζήτηση στο Συμβούλιο. Καταρχήν είδαμε τι έγινε στην Ιταλία. Ε, η Κομισιόν αντέδρασε άμεσα και ο κύριος Λάιτενεν θα μας το αναφέρει μετά για να συνδράμει τις Ιταλικές αρχές και γι' αυτό θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους Ιταλούς Επίσης η Frontex έχει ε, ανθρώπους δικούς της επιτόπου για να βοηθήσει την κατάσταση στη Λαμπεντούζα και η Europol επίσης δρά για να δει κατά πόσο υπάρχουν εγκληματικές δραστηριότητες. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις Ιταλικές αρχές για το ανθρωπιστικό τους έργο. Φαίνεται ότι η κατάσταση έχει κάπως καταλαγιάσει τα... τις τελευταίες ημέρες. Δεν έχουμε προσέλευση τηλησίων στη Λαμπεντούζα. Δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτή η τάση θα συνεχιστεί. Φαίνεται ότι πρόκειται για νέους τινήσιους με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που μπροστά σε αυτή τη χαοτική κατάσταση ήρθαν, προσήλθαν για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει διεθνής προστασία, αλλά φαίνεται ότι δεν έχουμε να κάνουμε με καθαρά οι οικονομικούς μετανάστες. Ως προς τη Λιβύη οι πληροφορίες αλλάζουν ώρα με την ώρα. Η κατάσταση είναι άκρος ανησυχητική. Είδαμε μία εκροή ανθρώπων προς γειτονικές χώρες, διότι όταν υπάρχουν τέτοιες σειράξεις, οι άνθρωποι προστρέχουν στις γειτονικές χώρες. χιλιάδες προς την Τινησία και την Αίγυπτο. Μερικοί είναι κάτοικοι Λιβύης που θέλουν να ξεφύγουν από αυτή την δραματική κατάσταση και μερικοί είναι την και Αιγύπτιοι. Αντιδράσαμε τάχιστα για να βοηθήσουμε αποστέλλοντας 3 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε στείλει ε, επιτόπου και δικούς μας ανθρώπους, η κυρία Γεωργίεβα είναι άκρος δραστήρια και ξέρουμε ότι η Υπάρχουν μεγάλες ανθρωπιστικές ανάγκες, ε, συνεργαζόμαστε με όλες τις αρχές για να έχουμε και τη δική τους εκτίμηση. Η Προεδρία μίλησε για το γεγονός ότι έχουμε 1.200 Ευρωπαίους πολίτες που προσπαθούμε να τους ε, βοηθήσουμε. Όταν μιλάμε για την κατάσταση ε, απόδρασης εκροών από τη Λιβύη, οι περισσότεροι δεν ήρθαν στην Ευρώπη, μετέβησαν στις γειτονικές χώρες, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι πολλοί θα προσέλθουν στην Ευρώπη. Θα δούμε τι θα γίνει στη Λιβύη. Δηλαδή, κατά πόσο πρόκειται για έναν εμφύλιο πόλεμο ευρεία κλίμακας, πώς θα... Ε, τι, τι, τι τέλος θα γνωρίσει η κατάσταση. Δεν έχουμε αριθμητικά στοιχεία, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενη κατάσταση. Γνωρίζουμε τι συνέβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοιτάξουμε και το θέμα της ε, κατεπίγουσας χρηματοδότησης. Έχουμε 25 εκατομμύρια ευρώ για περιπτώσεις επίγουσας ανάγκης. Θα πρέπει βεβαίως να προσβλέψουμε και σε άλλα μέσα, εκεί που χρειάζεται. Επίσης το Συμβούλιο μίλησε για την ενίσχυση της Frontex δηλαδή να προβάλλει νέα δράση με περισσότερο προσωπικό και εξοπλισμό, να δούμε κατά πόσο μπορούμε να διασφαλίσουμε την κατάσταση στη Μάλτα και την Ιταλία. Η ΙΑΖΟ δεν ε, έχει πλήρη δραστηριότητα στον τομέα του ασύλου, αλλά μπορεί να υποστηρίξει μερικώς τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να βοηθήσουμε στην ε, δράση έτσι ώστε να υπάρχουν υποδομές υποδοχής και επίσης να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μέσα διαθέτουμε. Θα πρέπει να μας απασχολήσει και η μακροπρόθεσμη υποστήριξη της κατάστασης. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική στον οικονομικό, κοινωνικό τομέα, στο τομέα της μετανάστευσης, στις γείτονες χώρες μας και είμαστε σε επαφή και με την IOM. Θέλουμε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε με έκτακτα μέτρα, όπως έγινε το Συμβούλιο, η Επιτροπή προσβλέπει σε νέα μέτρα, αλλά νομίζω ότι στο Συμβούλιο δεν ε, ελέγχθη κάτι άλλο με, την Επίτροπο, με, με τους Επιτρόπους Γεωργίευα Φίλε και με την ύπατη εκπρόσωπο Άστον καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να συνδράμουμε, αλλά η δραματική κατάσταση σημαίνει ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν ευθύνη μέσα στα πλαίσια μιας ευρύτερης αλληλεγγύης. Ε, λυπούμε που μακρηγόρησα, αλλά χρειάζομαι και το δικό σας input για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να συνδράμουμε στην κατάσταση. Ευχαριστούμε την Επίτροπο Μάλστρομ. Τώρα ο πρέσβης Μητήμων έχει το λόγο, που είναι ο Γενικός Γραμματέας της Frontex. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομο, γιατί νομίζω ότι τα περισσότερα έχουν ήδη υποθεί. Θα σας δώσω μόνο μερικές επιπλέον πληροφορίες, Ενδεχομένω μια διάκριση μεταξύ της Τινησίας και της Αιγύπτου από τη μία και της Λιβύης από την άλλη. Η κατάσταση όπως φαντάζεστε δεν είναι ακριβώς ίδια. Σε σχέση με τη Λιβύη, αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι μια τριπλή προσέγγιση. Πρώτον, η απομάκρυνση των Ευρωπαίων ε, υπηκών και θα ήθελα να επενέσω ιδιαίτερο στην Ουγγρική Προεδρία ε, ως προς αυτό γιατί πραγματικά ήταν πολύ εντυπωσιακό ε, το καθήκον που ανέλαβε σε πολύ δύσκολες συνθήκες και όπως σας είπε και η Επίτροπος αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου χιλίους, χίλιους Ευρωπαίους ακόμη στην περιοχή Και υπάρχουν μάλιστα και κάποιοι που δεν έχουν την πρόθεση να αποχωρήσουν. Το πρόβλημα που έχουμε και που θα έχουμε κατά τις ερχόμενες ημέρες ε, είναι πολίτες όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά από την Τινησία και την Αιγυπτό που ε, βρίσκονται στα σύνορα, συγκεντρώνονται στα σύνορα μεταξύ Τινησίας και Λιβύης και ζητούν βοήθεια για να επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους. Περίπου 20 με 30 χιλιάδες ε, Αιγυπτίους έχουμε αυτή τη στιγμή στην Τινησία και ε, θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους και η Αίγυπτος βέβαια κινητοποιεί τον εξοπλισμό της αλλά ζητεί την συνδρομή άλλων χωρών ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δεύτερη πτυχή και νομίζω ότι αυτό αυτή η πτυχή θα είναι όλο ένα και πιο εμφανής όσο περνούν οι μέρες, είναι η ανθρωπιστική συνδρομή. Γνωρίζετε ότι δεν ε, ε, μπορούσαν οι ανθρωπιστικές δυνάμεις να μπουν στη Λιβύη, στη Βεγγάζη και στο ανατολικό τμήμα κυρίως ε, της χώρας. Έχουν όμως, όταν πηγαίνουν βλέπουν μια εντελώς δραματική κατάσταση στα νοσοκομεία και προσπαθούν να βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο με φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό, ενδεχομένως και επισητιστική βοήθεια να χρειαστεί κατά τις ερχόμενες ημέρες. Όπως υπόθηκε και από την Προεδρία, Υπάρχει το όλο ζήτημα επίσης ε, της, ε, της ε, προσπάθειας καταστολής της βίας και επιβολής του νόμου στη Λιβύη. Οι κυρώσεις έχουν για την ώρα επιβληθεί και είναι πολύ εντυπωσιακό το πώς αποφασίστηκαν όλα αυτά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, είτε στη Νέα Υόρκη, είτε εδώ στις Βρυξέλλες. Λεπτό προς λεπτό παρακολουθούμε όλη την κατάσταση για να δούμε κατά πόσο πρέπει να ληφθούν νέα μέτρα. Ε, υπάρχει διεθνής ε, διαβούλευση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όσον αφορά την Αίγυπτο και την Τινησία, δύο πράγματα πρέπει να μας απασχολήσουν. Πρώτον, η πολιτική κατάσταση επειδή ε, υπάρχει ακόμη μεγάλη αβεβαιότητα κατά πόσο οι μεταβατικές προσωρινές αρχές προσπαθούν να τα καταφέρουν για τρία ζητήματα. Πρώτον, το θέμα τη συνταγματική μεταρρύθμισης, αναθεώρησης του συντάγματο. Δεύτερον, όσον αφορά το θέμα τη εγκαθίδρυσης ελεκλογική διαδικασία Και τρίτον, ε, κατά πόσο ε, θα πρέπει να γίνουν πρώτα βουλευτικέ ή προεδρικέ εκλογέ. Όλα αυτά είναι μεγάλα πολιτικά ζητήματα, σημαντικότατα, τα οποία συζητούνται αυτή τη στιγμή και στι δύο χώρε. Δεύτερον, η δεύτερη δράση που πρέπει να αναλάβουμε σε σχέση με αυτέ τι δύο χώρε είναι να δούμε και τις βραχυπρόθεσμες και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες τους στον τομέα, για παράδειγμα, της ε, οικονομικής ανάκαμψης και των κοινωνικών ε, ε, προβλημάτων. Ένα από τα ζητήματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε σύντομα είναι ειδικότερα αιτήματα από την Τινησία και την Αίγυπτο, ενδεχομένως αυτό να πάρει χρόνο, ε, τους έχουμε ενημερώσει για τη βοήθεια που μπορούμε να ε, τους ε, παρέχουμε και και προσπαθούμε να δούμε πώς ε, μπορούμε να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερο. Το ζήτημα τώρα είναι να υπάρχουν ειδικότερα αιτήματα από τη δική τους πλευρά, γιατί διαφορετικά θα βρεθούμε πάλι στην κατάσταση κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να επιβάλλει την ε, ε, συνδρομή της, ενώ θέλουμε να αποφύγουμε κάτι τέτοιο, θέλουμε να αποφύγουμε μια τέτοια στάση, γιατί ακριβώς αυτές οι χώρες αυτό δεν θέλουν πλέον. Θέλουμε ένα διάλογο λοιπόν επ' αυτού και θέλουμε να ε, συζητήσουμε, να συνεχίσουμε βάση διαλόγου. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνω στα πέντε λεπτά ακριβώς. Πέντε λεπτά ακριβώς και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Τώρα δίνουμε το λόγο στον ε, διευθύνοντα σύμβουλο της Frontex. Καλημέρα σας και εγώ θα πρέπει να είμαι ιδιαίτερα σύντομος. Έχω ετοιμάσει δύο διαφάνειες που ελπίζω να μπορέσετε να δείτε σύντομα. Όπως ε, προελέχθη, υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια ως προς την κατάσταση που επικρατεί. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα σενάρια που θα επικρατήσουν ποια σενάρια θα επικρατήσουν με βάση την παρούσα κατάσταση. Ε, επίσης, ο κύριος Βημού είπε πολύ σωστά ότι δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε αυτές τις χώρες ως μια ενιαία οντότητα. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές και γι' αυτό θα πρέπει να γίνει μια εκτίμηση χώρα προς χώρα. Αυτή είναι και η μόνη δυνατότητα. Ε, διαφορετικά σενάρια σημαίνει διαφορετικές μεταναστευτικές ε, ροές. Το θέμα της Τινησίας και το οποίο συνεχίζει να υφίσταται ως προς τη μετάβαση στη Λαμπετούσα είναι ένα παράδειγμα και όπως εξήγησε και η Επίτροπος είδαμε πως είχε η ε, σύνθεση αυτής της ε, ροής. Δηλαδή, είδαμε τι γίνεται όταν θα πρέπει να επιβληθεί ο νόμος. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο σενάριο όπου έχουμε να κάνουμε με μία μαζική ροή ανθρώπων οι οποίοι απεγνωσμένα προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο διαφυγής και το, το modus operandi, τα modi operandi είναι διαφορετικά ανάλογα με το σενάριο που επικρατεί. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι το εξής. Προσπαθήσαμε να αρχίσουμε με το, την επιχείρηση Ερμής μετά από αίτημα της Ιταλίας. Μπορέσαμε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα της Ιταλίας κατά 100% όταν πρόκειται για τεχνικό εξοπλισμό και προσωπικό. Βεβαίως, οι Ιταλικές αρχές προβαίνουν σε δραστηριότητες ε, screening, όχι μόνο στη Λαμπεντούζα που υπάρχουν 900 παράνομοι μετανάστες, αλλά και σε άλλους τόπους όπου οι Ιταλικές αρχές έχουν προβάλλει στέγη, έχουν παράσχει στέγη για αυτούς τους ανθρώπους. Μπορώ να σας πω ότι υπάρχει μια μονάδα ανάλυσης κινδύνου που λειτουργεί καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα απέστειλα μία επιστολή στα Ηνωμένα Έθνη στην Υπηρεσία για τους Πρόσφυγες και στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για να, συλλέξει στοιχεία, να συλλέξουν στοιχεία έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες από αυτές τις οργανώσεις θα ωφελήσουν και εμάς και τις δικές μας δραστηριότητες και αντιστρόφως. Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, με τη Europol, με την ΕΙΕΔ όπως σας είπα και όταν πρόκειται για το Γραφείο Υποστήριξης Μετανάστευσης έδωσα στους συναδέλφους όλα τα ε, διοικητικά στοιχεία υποστήριξης καθώς και επιχειρησιακή βοήθεια. Ορισμένα στοιχεία ως προς την επιχείρηση Ερμής. Όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή έχει τεθεί σε λειτουργία και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τι θα γίνει μετά από τι έγινε μετά τις 26 Φεβρουαρίου που δεν είχαμε νέα προσέλευση. Φαίνεται ότι οι αρχές της ε, Τινησίας είναι ιδιαίτερα δραστήριες και μετά από αυτή τη βραχή περίοδο που δεν ήταν δραστήριες οι αρχές μπόρεσαν να ανταποκριθούν. Ο συνολικός αριθμός βλέπετε στις μεγάλες φούσκες εκεί, η πράσινη αφορά τις αρχές διευκόλυνσης και το μπλε είναι τα επεισόδια που γνωρίσαμε εκεί όπου έφτασαν οι παράνομοι μετανάστευς. μετανάστες. Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε με βάση το επιχειρησιακό πακέτο. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε τον δικό μας εξοπλισμό και προσωπικό, γι' αυτό η διαδικασία είναι κάπως χρονοβόρα. Θα πρέπει να έχουμε μια ιδιαίτερα δραστήρια προσέγγιση και να μην υπάρχουν οικοτολογίες, πανικός και όλα τα σχετικά. Η Μάλτα, όπως γνωρίζουμε, υφίσταται μεγάλη πίεση και χρειάζεται βοήθεια από τα άλλα κράτη-μέλη και Σήμερα το βράδυ θα μεταβώ στη Μάλτα για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να επεκτείνουμε την επιχείρηση Ερμής. Τέλος, θα ήθελα να μιλήσω για την Ελλάδα. αν και φαίνεται ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο στα ελληνοτουρκικά σύνορα και έχουμε μείωση κατά 75% ε, ροών σε σχέση με τις αρχές Νοεμβρίου, η κατάσταση είναι αρκετά απαιτητική και δεν μπορεί να διαχωριστεί από το τι συμβαίνει στη Βόρειο Αφρική. Γιατί ότι οι πτήσεις ήταν από το Μαγκρέμπ στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια μετέβαιναν οι μετανάστες αυτοί προς την Ελλάδα. Και χρησιμοποιήθηκε αυτή η οδός προς την Ελλάδα από μετανάστες από τις χώρες ε, του Μαγκρέμπ. Όπως ανέφερε και η Επίτροπος, εάν θα πρέπει να, να συνεχιστεί αυτή η περίοδος ε, πήγουσας ανάγκης, θα πρέπει να προστρέξω στις αρχές προϋπολογισμού για επιπρόσθετο προϋπολογισμό και προσωπικό. Ευχαριστούμε κύριε Λατίνεν. Τώρα θα έχουμε ένα πρώτο γύρο ε, παρεμβάσεων από τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων και μετά προτείνω να ακούσουμε από τον εισηγητή για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Λιβύης από την κυρία Άννα Γκόμες και από την αντιπροσωπεία από τον κύριο Πανζέρη που είναι ο πρόεδρος της Μικτής Επιτροπής ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών Μαγκρέπ. Προτείνω λοιπόν ο καθένας, ο κάθε συντονιστής να αρκεστεί σε δύο 25 λεπτά έτσι ώστε να τα καταφέρω. Η κυρία Μόρβαϊ. Το συνήθως ερώτημα. Τα μία για μέλη παρακαλώ να έχουν επίσης δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις. Μα οπωσδήποτε, στο δεύτερο γύρο θα μπορείτε να μιλήσετε. Πρώτα θα ακούσουμε τους συντονιστές. Ο κύριος ο πρώτας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν όλους τους MDs ε, που ήρθαν εδώ, δέχτηκαν την πρόσκλησή μας και μας έκαναν την παρουσίασή τους. Ομολογώ ότι με ενθαρρύναν αυτά που άκουσα, γιατί είναι προφανώς ε, έχουν την κατάσταση υπό έλεγχο. Αυτό είναι πολύ καλό. Η κατάσταση είναι πολύ θετική. Εγώ είμαι από τη Μάλτα και σε μια εβδομάδα, μόνο την περασμένη εβδομάδα, η χώρα μου ε, 12.000 προσφύγους από τη Λιβύα από 89 διαφορετικές χώρες. 12.000, επαναλαμβάνω. Το γεγονός ότι όλα αυτά έγιναν ομαλά οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι είχαμε διάφορα κράτη-μέλη, διάφορα χώρες που έστεναν αεροπλάνα για να πάρουν τους δικούς τους υπηκόους. Τι θα γινόταν αν οι 12.000 αυτοί ήταν Λίβοι, θα είχε στείλει κανένα αεροπλάνο για να βοηθήσει. Ελπίζω ναι. Ποιε είναι οι προτεραιότητε μα. Η πρώτη προτεραιότητα είναι σαφή. Θα πρέπει να σταματήσει η βία. Αυτό θα πρέπει να είναι η πρώτη μα και πολύ σαφή μέρημνα. Χαιρετίζω την εισαγωγή των κοινοτικών κυρώσεων, παρόλο που φοβούμαι ότι δεν θα αρκέσουν να σταματήσουν τη βία αυτή τη στιγμή. Η δεύτερη σαφή μα προτεραιότητα είναι να αποστείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της Λιβύης. Είναι σαφές ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πια τρόφιμα, δεν έχουν φαρμακευτικά διασκευάσματα και θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να τους αποστείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Η τρίτη προτεραιότητα, τρίτη κατά τη γνώμη μου, είναι ε, τι θα κάνουμε για το ενδεχόμενο μεταναστευτικό κατεπήγον που θα δημιουργηθεί. Προφανώς κανένας δεν το θέλει, αλλά ίσως λάβει χώρα, όπως έγινε και μεταξύ Λιβύης, Ισίας και Αιγύπτου. Και πιστεύω ότι αυτές οι, οι ζώνες είναι ήδη ζώνες ε, ανθρωπιστικής κατεπίγουσας ανάγκης. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια σαφή απάντηση τι θα γινόταν δηλαδή εάν έχουμε μαζική ροή από τη Λιβύη προς την Ευρώπη. Είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε. Τι θα κάνουμε. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε χιλιάδες ατόμων που φεύγουν από την Λιβύη προς την Ευρώπη. Υπάρχει ένα σχέδιο Frontex έτοιμο για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί αν λάβει χώρα κάτι τέτοιο. Και αυτοί τους οποίους θα βοηθήσει η Frontex να φύγουν από τη Λιβύη, πού θα πάνε στα απελευθερωμένα τμήματα της ε, Λιβύης, στην περιοχή της Μπενγκάζη ή σε διάφορα καρδιμέλη. Και αν ναι, ποια. Ξέρω ότι όπως είπε και η κυρία Μάστρομ στο Συμβούλιο δεν υπάρχει φαίνεται κανένα ενδιαφέρον για να υποδεχθούν τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη κατάσταση και θα πρέπει για μια δύσκολη κατάσταση να είμαι έτοιμη να την αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Ο κύριο Μωράη, δύο μισή λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Νομίζω το έργο που έχουν εκτελέσει οι ε, προσκεκριμένοι μας σήμερα είναι πραγματικά πολύ εξεπρόσευτο. Το Κοινοβούλιο, και δεν πρέπει να ξεχνάμε το Κοινοβούλιο έχει επισκεφθεί τη Λιβύη, έχει κατ τα, να καταλάβει τα προβλήματα μετανάστευσης και προσφύγων στη Λιβύη με στα πλαίσια της Frontex. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πίεση στη Μάλτα, τίποτα το καινούργιο εκεί. Το γεγονό ότι στην Λαμπεντούσα δεν υπάρχουν πια την ίση πρόσφυγες, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω στα συμπεράσματα του Συμβουλίου ελέγχθη ότι δεν ενδιαφέρεται κανένας να μεταφέρει αυτούς τους ανθρώπους στην Ευρώπη και ενδεχομένω για να υπάρχει κατανομή των βαρών. Έχουμε όμως το πρόβλημα αυτό. Η επίγουσα κατάσταση στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Μπουζουτήλ είναι σημερινή κατάσταση. Πολλοί από εκείνους που πήγαν στην Λαμπεντούζα από την Ισία είναι άνθρωποι με πανεπιστημική μόρφωση. Είναι άνθρωποι που θα έρθουν στην Ευρώπη τελικά και δεν πρέπει να προσποιούμε ότι δεν θα έρθουν, θα έρθουν. Λοιπόν, Ρωτάω, υπήρχε μια αίσθηση κατεπήγοντα στο Συμβούλιο την Παρασκευή που έλεγε ότι δεν θα έχουμε έτοιμα τα νέα μέσα για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της κατανομής του βάρους, τις διαδικασίες, όλα αυτά έχουν καθυστερήσει στο ίδιο το Συμβούλιο που προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα. Δεν είναι θέμα της Κομισιόν αυτό. Σας ρωτάω λοιπόν, είχατε την ότι έχουν στην αίσθηση του κατεπήγοντος. Και δεύτερη ερώτηση, αν υπάρχει σχέση του κατεπήγοντος, δεν θα πρέπει να μιλήσουμε μεσοπρόθεσμα κάποια στενή εταιρική σχέση με τις χώρες πρόλευσης που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όπως υπάρχει μεταξύ Λιβύης και Ιταλίας, παραδείγματος χάρη, αλλά πραγματικές εταιρικέ σχέσεις που λαμβάνουν υπόψη τις ε, μόνιμες αλλαγές ε, της φύσης των σχέσεων των χώρων αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολλοί νέοι, καλά εκπαιδευμένοι, που θα έρθουν εδώ δεν υπάρχει καμία έννοια να έχουμε έτσι γενικέ και όριστε ιδέε για την κατανομή του βάρου. Και αυτά που είπε ο κ. Μπουζουτέλ για τη Μάλτα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Η ομάδα μου αναρωτιέται λοιπόν, ξέροντα τα προβλήματα αυτά, θα υπάρχει κατεπίγουσα προσπάθεια του Συμβουλίου για το, την οδηγία για το άσυλο, για τη μετανάστευση. Και συζητάμε τώρα για τον περιορισμό της κρίσης ή για μεσοπρόθεσμες και, και μακροπρόθεσμες λύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βέμπερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους διακεκριμένους επισκέπτες που ήρθαν εδώ σήμερα. Θα σας ευχαριστήσω που ήρθανε, που μας έκαναν τις παρουσιάσεις τους και πραγματικά ότι ανέτρασαν τόσο σύντομα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας νομίζω, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να είμαστε ενημεροί, να έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλουμε ερωτήσεις και να διευκρινίσουμε κάποια θέματα. Προσωπικά θα ήθελα να μου τρέψει να σας πω ότι προφανώς το 1989-1990 όταν έγιναν οι αλλαγές στον καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ήταν ανέτοιμες και βέβαια δεν είναι εξεπλαγμένο ότι και τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν και πολύ έτοιμη για τις αλλαγές αυτές του καθεστώτος στην Βόρεια Αφρική. Καταλαβαίνω βέβαια και είναι σαφές ότι θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ των, στην αφενός και της Λιβύης αφετέρου και ποιος ξέρει και ποιες άλλες χώρες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Είμαστε λογικοί άνθρωποι βέβαια και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και εκεί Ευρωπαίοι επίκοοι που αποτελούν την προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα όμως το χειρότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς σκοτώνονται άνθρωποι στη Λιβύνη. πεθαίνουν άνθρωποι εκεί και αυτό για αρκετό καιρό τώρα. Και υπάρχουν φωνές όχι μόνο οι δικοί μου που λένε ότι «Ε, και αυτή τη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντέδρασε όποτε θα έπρεπε να έχει αντιδράσει. Λίγα πράγματα, όχι πολύ έντονα. Καταλαβαίνω βέβαια ότι τώρα προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Έχω μια-δυο ερωτήσεις. Από ό,τι κατάλαβα, η Frontex ήδη εργάζεται βάσει διαφορετικών σεναρίων ανάλογα τι θα έχει γίνει, τι θα γίνει, έχουν τους ε, η εμπειρογνώμας ανάλυσης και καταλαβαίνω ότι σε επίπεδο Κομισιόν έχετε αυτήν τη συνεργασία που έχετε. Αλλά ρωτάω, ίσως θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο κύτταρο κρίσης που μπορεί να κινητοποιηθεί κάθε φορά που χρειάζεται και να εργαστεί η βάση προγραμμάτων ΑΒΓ. Γιατί αυτό θα ήταν για μας πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν θα αφορούσε μόνο τη δράση, αλλά και το θέμα των, ε, των πόρων ένα ταμείο κατεπίκουσας βοήθεια 25 εκατομμυρίων. Δεν τίποτα αν η Λιβύη είναι όπως είναι. Ευχαριστώ κύριε Σαγεντίνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν κάποιος φεύγει από μια χώρα που δεν ε, είναι ασφαλής, είναι πρόσφυγας και επομένως είναι κοινικό να λέμε ότι στέλνουμε πλοία και αεροπλάνα για να, για να, για να ε, ε, φύγουν οι Ευρωπαίοι πολίτες από εκεί. αναρωτιέμαι κατά πόσο ο εκπρόσωπος της Frontex ε, ή ε, η Επίτροπος μπορεί να μας πει τι γίνεται με τις συμφωνίες μεταξύ Ιταλίας και Λιβύης ε, και των συμφωνιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λιβύης. Ποιος κάνει περιπόλους τώρα στη Μεσόγειο για να ξέρουμε πώς ακριβώς ε, γίνονται μετακινήσεις. Και επίσης ο εκπρόσωπος της Frontex μας είπε ορισμένα πράγματα για την παρακολούθηση των μεταναστών, ε, το screening στην Ιταλία. Γιατί όταν είχαμε πάει στην Αθήνα, είχαμε καταλάβει ότι ένας πρόσφυγας δεν μπορούσε να ζητήσει άσυλο σε ένα συγκεκριμένο ε, συνοριοφύλακα της Frontex ε, και γι' αυτό αναρωτιέμαι τι ακριβώς είναι το screening, ε, από ποιον γίνεται και επίση πόσε αιτήσει για άσυλο έχουμε ε, μέχρι τώρα από τις χώρες Μαγκρέμπ. Επίσης, Έχουμε ξεχάσει ότι πριν από τις καλοκαιρινέ διακοπές μιλούσαμε εδώ για όσους είχαν καθυλωθεί στην ε, ε, έρημο και υπήρχε περίπτωση να επιστρέψουν στην Ερυθρέα και ποιες ήταν ε, οι συμφωνίες που είχαμε με τη Λιβύη ε, επ' αυτού. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν μια νέα αξιολόγηση των ανθρώπων με τους οποίους συναλλασσόμαστε και να δούμε πώς μπορούμε να ε, να μην ε, μεταφέρουμε τις δικές μας ευθύνες σε άλλους. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ε, ότι αυτοί οι άνθρωποι που καθαρίζουν από τους μετανάστες στη Μεσόγειο είναι αυτοί οι οποίοι καταπιέζουν τους λαούς τους. Όσον αφορά τώρα τη Λαμπεντούζα, δεν υπάρχει πια εισρωή μεταναστών γιατί οι Λίβοι έκαναν τόσο καλή δουλειά αστυνομεύοντας τη Μεσόγειο. Αυτό είναι πάρα πολύ κοινικό να το πει κανείς. Και μία ακόμη και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Μωράε από τους Σοσιαλδημοκράτε ότι θα έπρεπε να το δούμε ως προσωρινή κρίση αλλά πρέπει να βρούμε και μια πραγματική λύση και χρειάζεται το Συμβούλιο οπωσδήποτε τις πολιτικές μετανάστευση και ασύλου επιτέλους να τη βάλει σε τάξη. Δεν βλέπω τον κύριο Κίκοπφ εδώ για την ομάδα συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Οπότε ο κύριος Σταβάρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ε, ε, πληροφορίες ε, σε σχέση με το τι προγραμματίζουμε. Από ό,τι κατάλαβα εγώ, πρόκειται για μια τεράστια επιχείρηση συνόρων, εποπτεία συνόρων, επίβλεψη συνόρων, πολύ μεγάλης κλίμακας. Τι θα γίνει όμως αν ε, είναι μια τεράστια ε, ανθρωπιστική επιχείρηση. Μπορεί μια εποπτεία των συνόρων να μην επαρκεί. Έχουμε 5.000 χιλιόμετρα από το Μαρόκο στη Συρία. Υπάρχει τεράστια ανθρωπιστική απειλή στην περιοχή και δεν με ανακουφίζει καθόλου το γεγονός ότι ε, είναι διαφορετικές οι χώρες όπως είπε ο κύριος Βιμόντ Μπορεί να έχουμε 10 διαφορετικέ καταστάσει. Αλλιώ είναι η κατάσταση στα σύνορα Μαρόκου-Αλγερία, αλλιώ ε, είναι η κατάσταση στα σύνορα Συρία και Τουρκία, όπου υπάρχουν ακόμη πρόσφυγε από το Ιράκ. Οπότε, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ποιο είναι, ποιος είναι ο δικό μα βαθμό ετοιμότητα στα δικά μα σύνορα σε σχέση με τη δική μα ικανότητα να επεξεργαστούμε αυξημένε αιτήσει ασύλου και ειδικότερα σε σχέση με την αλληλεγγύη για ε, την. Ε, για τον επαναπατρισμό. Γιατί υπάρχει μεγάλη σύγχυση μεταξύ μεταναστών και ε, τούντων άσυλο, ειδικότερα στην περίπτωση της ε, Τινησίας. Ε, το είπαμε και στο Στρασβούργο αυτό. Στην Τινησία υπάρχει ένας νόμος, όταν γυρίσει ένας μετανάστης πίσω στην Τινησία, είναι ένας εγκληματίας. Οπότε πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια αυξημένη εισρωή ετούντων άσυλο. Εμείς στη συναπόφαση μας ε, είχαμε προβλέψει το, το εξής. Πρώτον, είχαμε πει ότι υπάρχουν κάποιες ε, περιοχές προτεραιότητας, κατεπίγουσας προτεραιότητας. Ε, το είχαμε συζητήσει, το έχουμε συζητήσει και σε τέτοιου είδους συνεδριάσεις πολλές φορές. Οι ανθρωπιστικές κρίσεις δεν έχουν ημερομηνία, μπορεί να γίνει ε, κάτι το Φεβρουάριο ή το Μάρτιο και να πρέπει να μεταφέρουμε τις προτεραιότητές μας από τις χώρες του Μαγκρέπ στις χώρες του Μασρέπ, για παράδειγμα. Ε, επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα που ανέφερε και η Ρενάτα Βέμπερ ε, για ένα, μια ομάδα ε, κρίσης σε, περίπτωση τέτοιων, κρίσεων. Αυτό που με απασχολεί επίσης είναι ο βαθμός ε, εξάρτησης που έχουμε από δικτάτορες ε, για να δούμε τις δικές μας μη ρεαλιστικές μεταναστευτικές πολιτικές. Πρέπει να το σκεφτούμε. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας είπε ότι ε, δεν έχει καταργηθεί, δεν έχει καταπέσει η Συμφωνία Ιταλίας και Λιβύης, απλώς de facto δεν είναι επιχειρησιακή τι θα κάνουμε όμως. Πρέπει να είμαστε κι εμείς αξιόπιστοι, πρέπει να, ε, έχουμε συγκεκριμένα, ε, συγκεκριμένες πολιτικές τις οποίες οι, πολιτικοί, οι πολίτες μας μπορούν όντως να έχουν εμπιστοσύνη. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω, λέει ο κύριος Μποργέζιο, τους προλαλήσαντες και τους ηθήνοντες που μας δώσαν ε, πολλές πληροφορίες, θα ήθελα να ρωτήσω ποια θεωρούνται επαρκή κριτήρια. Μιλάμε για 25 εκατομμύρια ευρώ. Δεν αρκούν. Δεν αρκούν αν λάβουμε υπόψη το τι συνέβη που είχε τεράστιες διαστάσεις όχι μόνο στη Μάλτα, αλλά και στη Λαμπεντούζα. Πρόκειται για μία κατάσταση επίγουσας ανάγκης και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την στάση των κατοίκων της Λαμπεντούζα που ήταν εξαιρετική, δηλαδή υποδέχτηκαν ε, τους μετανάστες χωρίς να, έχουν ε, τάση, να δείχνουν κάποια τάση να τους αποδιώξουν, χωρίς να έχουν ε, τίποτα να προσφέρουν επί της ουσίας, αρχίζοντας και από την κατάσταση υγείας και υγειονομικής. Αυτό, θα πρέπει να λάβουν, αυτό που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι υπάρχουν πολλά κενά στην πολιτική μας διότι αυτές οι, οι μεταβάσεις δεν ε, έχουν προσλάβει μεγάλες διαστάσεις αυτές οι μέρες διότι υπάρχει μεγάλη θαλασσοταραχή στην ε, περιοχή. Όταν θα κοπάσει η θαλασσοταραχή τότε ε, θα υπάρξουν αυτές οι εκροές. Και θα δούμε τι θα γίνει όταν θα σκάσει και η φούσκα της Λιβύης. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ποια μέτρα θα αναλυφθούν για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την κατάσταση επίγουσας ανάγκης. Δεν έγινε καμία μνήμα σε αυτό. Καθίσταται σαφές ότι οι χώρες όπως η Μάλτα και η Ιταλία δεν μπορούν να αφαιθούν στην τύχη τους. Άκουσα πολλά για αλληλεγγύη. Έγινε λόγος για τη Σουηδία, για το Βέλγιο, που είπαν ότι σε μια κατάσταση επίγουσας ανάγκης δεν θα δεχτούν ούτε έναν μετανάστη. Αυτό μας είπαν αυτές οι δύο χώρες. Γι' αυτό θα ήθελα να ξέρω πώς θα γίνει μια σωστή κατανομή για να μπορέσουμε υπεύθυνα να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Αυτό είναι ένας ε, γόρδιος δεσμός, τον οποίο θα πρέπει να ε, λύσουμε και όχι βία, γιατί δεν μπορείτε να αφήσετε τη Μάλτα και την Ιταλία στην τύχη τους. Θα ήθελα επίσης να μου πει επίτροπος ε, τι σκέφτεται για την πρόταση Μαρόνι του Υπουργού Εξωτερικών της Ιταλίας Μαρόνι για ένα νέο σχέδιο Μάρσαλ γιατί αν δεν μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες in situ, δεν θα είμαστε σε θέση να μιλήσουμε για μια σοβαρή πολιτική μετανάστευσης. Βλέπω ότι η συνάδελφος Άννα Γκόμες, που είναι η συγγήτρια για την έκθεση ως προς την κατάσταση στη Λιβύη, δεν είναι παρούσα πλέον. Γι' αυτό θα ακούσουμε από τον κύριο Παντζέρη που είναι πρόεδρος Μικτής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Χωρών Μαγκρέμπ και μετά θα γίνει συζήτηση με τα μέλη. Ο κύριος Παντζέρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Γνωρίζουμε ότι οι μεταβάσεις, οι μεταβατικές καταστάσεις δεν είναι εύκολες όπως μας καταδείκνει η Τινησία και η Αίγυπτος. Η Τινησία και η Αίγυπτος και η κατάσταση στη Λιβύη είναι ακόμα πιο δυσχερής. Πρόκειται για μια διαδικασία που δεν θα γνωρίσει τέλος το εγγύς μέλλον. Γι' αυτό θα πρέπει πάντα να λάβουμε υπόψη αυτές τις πτυχές του ζητήματος. Δηλαδή οι δύο επίτροποι Μάλστρομ και Φίλε θα πρέπει να, είναι σε, να βρίσκονται σε στενή συνεργασία. Οι άμεσες δράσεις ήταν πολύ καλές, η επιχειρησιακή βοήθεια, αλλά θα πρέπει να έχουμε έναν μεγάλο ορίζοντα εάν λάβουμε υπόψη ότι οι μετανάστες δεν θα σταματήσουν στα όρια, στα σύνορα της Τινησίας. Θα μεταβούν πέραν της Τινησίας. Γι' αυτό θα ήθελα η Επίτροπος άμεσα να θέσει επιτάπητος την αύξηση πόρων, γιατί 25 εκατομμύρια δεν αρκούν πλέον. Είναι ε, ένα μελιτέο ποσό. Θα πρέπει επίσης να γίνει μια σωστή επανακατανομή του θέματος. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το θέμα εντασσόμενο μέσα σε μία γενικότερη στρατηγική. Και η στάση των ΙΠΑ θα πρέπει να μας καταδείξει ότι θα πρέπει να δράσουμε επιτόπου και άμεσα. Και μακροπρόθεσμα βεβαίως. Συμφωνούμε ότι η Επιτροπή Γειτονίας και Εταιρικότητας θα πρέπει να κινηθεί προς νότον μέσα στα πλαίσια της εθνικής κυριαρχίας. Και θα ήθελα να πω προς τον Δόκτρα Βήμο ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στην Ισία άμεσα, διότι θα είναι ένα σημείο αναφοράς, έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε την δημοκρατική διαδικασία και θα πρέπει να υποστηρίξουμε όχι μόνο την δημοκρατική διαδικασία, αλλά να προωθήσουμε επί τόπου τάχιστες δράσεις. Διότι θα είναι η πρώτη χώρα η Τινησία η οποία θα οδεύσει προς τη δημοκρατία. Τώρα προσήλθε η Άννα Γκόμες και έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον πρέσβη κύριο Βήμα που αναφέρει ότι η προτεραιότητα είναι να σταματήσει η, η βία και η επίτροπος μάλιστα με το ίδιο. Καλό να σταματήσει η βία. Να σταματήσουμε... Did nothing all these years. Ξέρουμε ότι ένας ψυχοπαθής, ε, ο ψυχοπαθής μάλλον που είναι στην ε, ε, εξουσία, έχει και πυρνικά όπλα. Γιατί να μην πούμε, εντάξει, δεν έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για κάτι τέτοιο. Σκεφτόμαστε ποιες θα είναι οι άλλες επιλογές που θα υπάρχουν επί τόπου, όπως είπαν οι Αμερικανοί. Ιδίως γιατί έχουμε την ευθύνη να προστατεύσουμε τους ε, Λίβιους πολίτες και όποιους μετανάστες έχουμε την υποχρέωση να προστασέψουμε στις 100.000 Ευρωπαίους πολίτες που είναι εκεί. Δεύτερο, τι γίνεται με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Ποια είναι η ευρωπαϊκή μας προτεραιότητα. Να κρατήσουμε εκτός Ευρώπης αυτές τις ορδές και να χρησιμοποιήσουμε τη Frontex για να τόσο αποκλείσουν ή θα πρέπει να υπάρχει μια πραγματική πρόθεση ανθρωπιστικής βοήθειας που όχι θα μας δώσει οραματικότητα που δεν έχουμε. Κοιτάξτε, ό, σε οποιοδήποτε σταθμό της τηλεόρασης θέλετε, ούτε στην ε, Τουνησία, ούτε στην Αίγυπτο, ούτε πουθενά. Και δώνοντας αυτή την ανθρωπική βοήθεια, διευκολύνοντας την, είπα το αρμοστία για τους πρόφυγες του ΙΕ, δεν θα ήταν αυτός ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς και να τους αποκλείσουμε από το να έρθουν εδώ, όχι να τους απογρεύσουμε να του βοηθήσουμε επί τόπου. Δεύτερον, υπάρχουν πολλοί ε, μετανάστες που δεν είναι ούτε Αιγυπτιού ούτε Ινωσία, το Σουδάν από την Ερυθρέα, οι πιο ευάλωτοι είναι αυτοί, οι πιο φτωχοί. Τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θα πρέπει γι' αυτό να έχουμε εκεί την υπατιαρμοστία ε, ε, να δράσουν ιδίως στην ε, περιοχή της Μπεγκάζη. Τελευταίο ερώτημα οι κοινωτικές προσπάθειες για επίδραση στους νέους πολιτικούς δράσεις που θα διαδεχθούν αυτό το στρογαθή. Τι γίνεται με την ενθάρρυνση των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τι κάνουμε για να επιδράσουμε πολιτικά στη νέα, στο νέο καθεστώς που θα δημιουργηθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκόμες πρώτο γύρο αντιδράσεων με την ίδια σειρά όπως το πρώτο γύρο. Ο πρέσβης Κιόρκος είναι ο πρώτος που εκπροσωπεί την Ουγγρική Προεδρία. Παρακαλώ, έστε σύντομος κατά το δυνατόν. Uh, uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την αναγνώριση ε, όσον αφορά την αναγνώριση των προσπαθειών που έκαναν οι, ε, οι υπηρεσίε μας. Ε, ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά ήταν μια ερωική προσπάθεια. Όσον αφορά τώρα τον καταμερισμό του βάρους, θα ήθελα να σας ευχηστήσω την προσοχή στο, στο ότι Υπάρχει τεράστιος όγκος προσφύγων ε, που ε, έφτασε στην Ευρώπη και το 2010, οπότε υποθέτω ότι Πρέπει να λάβουμε υπόψη την κατάσταση αυτή όταν βλέπουμε τον οριζόντιο καταμερισμό βάρους ε, μεταξύ των χωρών. Όσον αφορά τώρα το πακέτο του ασύλου και της μετανάστευσης, είναι πραγματικά μία ένδειξη του κατά πόσο σοβαρά παίρνει το ζήτημα αυτό ε, της, ε, του θέματος της Βορείου Αφρικής. Είναι στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου. Το πακέτο ασύλου και μετανάστευσης θα είναι επίση πάρα πολύ σημαντική προτεραιότητα και τον Ιούνιο. Γνωρίζετε ότι έχουμε ήδη προς, ξεκινήσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες και θα τι εντείνουμε επόμενες εβδομάδες, εβδομάδε. Θέλουμε όσο το δυνατόν το κοινό σύστημα ασύλου ε, συντομότερα να το ολοκληρώσουμε. Το ζήτημα τώρα των ε, επιπτώσεων ε, της μη εφαρμογής ε, Συμφωνίας Ιταλίας-Λιβύης πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι για την ώρα οι μεταναστευτικές ροές στην Λιβύη, μεταξύ Λιβύης και Αιγύπτου και την Ισίας, κινούνται οριζοντίως, σε οριζόντια κλίμακα. Αν υπάρξει τώρα μια κάθετη τάση, θα είναι τεράστια πρόκληση για την Ευρώπη, αλλά όπως είπα υπήρξε μεγάλη μεγάλη πίεση ε, προς τα κράτη-μέλη και στις ε, αρμόδιες αρχές. Θα τα ακούσουμε άλλωστε και από τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Frontex, της Frontex, γιατί είναι σε θέση να ελέγξουν την κατάσταση και να προετοιμαστούν αν υπάρξει ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ. Η Επίτροπος Μάλμστρομ. Ευχαριστώ πολύ πρέπει οπωσδήποτε αμέσως να βοηθήσουμε τις ε, ε, γειτονικές της Λιβύης χώρες για να αντιμετωπίσουν αυτή την ανθρωπιστική κατάσταση, ε, την ανθρωπιστική κρίση. Οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι παρούσες επιτόπου, αποστέλλονται κονδύλια, ανθρωπιστικός εξοπλισμός και ε, βέβαια παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό την κατάσταση. Δεν υπάρχει επίσημη ομάδα κρίσης, υπάρχει όμως ανεπίσημη. Εγώ είμαι σε ημερήσια βάση σε επαφή με την ε, με τον κύριο Φίλε, με την κυρία Γεωργίευα, με την Προεδρία, ε, με όλους όσους συμμετέχουν στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης αυτής. Υπάρχει λοιπόν μία ομάδα, ο κύριος Γκουτέρες για παράδειγμα συμμετέχει σε αυτή την ομάδα ε, για ε, την παρακολούθηση της κατάστασης. θα, θα ήταν πολύ καλό βέβαια να έχουμε ήδη το κοινό σύστημα ασύλου αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι μια μεγάλη μας επιθυμία και είμαι σίγουρη ότι η Ουγγρική Προεδρία κάνει ό,τι μπορεί για να προχωρήσει το θέμα αυτό και μπορώ μόνο να ενθαρρύνω τα κράτη-μέλη να το πράξουν ε, και εκείνα. Βλέπουμε τα διάφορα σενάρια που κινούμε τη Frontex και τα διάφορα κέντρα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 αιτήσεων ασύλου. Μίλησα για 25 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στη διάθεση της ε, αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι, δεν είναι επαρκή, πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε περισσότερους πόρους, να εντοπίσουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Ε, έχουμε και το άρθρο 78 εδάφιο 3 που μας δίνει τη δυνατότητα να αντλήσουμε πόρους προκειμένου να υπάρξουν επιπρόσθετα να υπάρξει επιπρόσθετη χρηματοδότηση για τέτοιου είδους περιπτώσεις. Όλα αυτά τα έχουμε ήδη δρομολογήσει και προσπαθούμε να δούμε και τις διάφορες δυνατότητες που έχουμε να βοηθήσουμε και σε ανθρωπιστικό επίπεδο. Όπως είπε και ο κύριος Μπουσούτιλ και άλλοι, μιλήσατε για την όρεξη ε, εσωτερικής μετεγκατάστασης ε, των ε, μετακίνησης των μεταναστών. Δεν είναι τεράστια αυτή η όρεξη. Είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Θέλουμε να βοηθήσουμε. Προσπαθούμε να συζητήσουμε και με τον κύριο Λάιτινεν να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να βοηθήσουμε βοηθήσουμε τον, τα κράτη-μέλη. Είμαι σίγουρη βέβαια ότι η Μάλτα βρίσκεται υπό ιδιαίτερη πίεση και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξουν πολλέ ε, προσπάθειες από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπάρχει βέβαια και μακροχρόνια προοπτική να βοηθηθούν οι χώρες αυτές. Πρέπει να συμπεριλάβουμε μέτρα νόμιμη ε, νόμιμης Αυτό όμως είναι μια μακροχρόνια προοπτική και το επεξεργαζόμαστε από κοινού με την, την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Οπότε νομίζω ότι Αυτά που μπορούμε να κάνουμε τα κάνουμε ήδη και εξετάζουμε τα διάφορα σενάρια. Ακόμη και αν ε, δεν έχουν φτάσει ακόμη οι άνθρωποι αυτοί στην Ευρώπη, κάποια στιγμή θα φτάσουμε και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Δεν υπάρχει καν, καμία ε, περίπτωση να στείλουμε πίσω ανθρώπους που έχουν ανάγκη ε, βοήθειας. Υπάρχουν διεθνείς νόμοι για τα ζητήματα αυτά, του οποίου πρέπει να σεβαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο γενικό Γραμματέας Βημό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που ελέγχθησαν από την Επίτροπο και τον εκπρόσωπο της Προεδρίας του Συμβουλίου. Εξετάζοντας τα δεδομένα, θα πρέπει νομίζω να κάνουμε μία διάκριση μεταξύ της, των διαφόρων ε, τύπων μεταναστών εντό εισαγωγικών που βλέπουμε. Καταρχήν έχουμε τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί ή θέλουν να πάνε στις πατρίδες τους. Μετά έχουμε τους Τινησίους και τους Αιγυπτίους πολίτες που επίσης περνάνε τα σύνορα για να πάνε σπίτια τους. Το πρόβλημα, ένα από τα προβλήματα που έχουμε είναι στα νησιακά σύνορα είναι ότι έχουμε παραδείγματος στους Αιγυπτίους που θέλουν να πάνε στην ε, πατρίδα τους και θα υπάρχει και μια διάκριση όπως το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Στα σύνορα μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης ο Αιγυπτιακός στρατός ασχολείται με τα πάντα και εργάζεται με μεγάλη τάξη από ό,τι βλέπουμε. Τα πράγματα προχωράνε πολύ καλά. Στα σύνορα με την Τινησία υπάρχει μια έλλειψη ανθρωπίνων πόρων, αν θέλετε, και εξοπλισμού και εκεί υπάρχουν οι αιτήσει βοήθειας από την διεθνή κοινότητα. Και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια άλλη ομάδα που δεν έχει αναφέρει κανένας. Είναι οι πολίτες τρίτων χωρών. 25.000 Κινέζοι, παραδείγματος χάρη, εξίσου Τούρκοι, άνθρωποι από τις Φιλιππίνες που ζητάνε βοήθεια. Και αυτούς προσπαθούμε επίσης να βοηθήσουμε για να τους ε, πάμε στις ε, χώρες τους παραδείγματο χάρη είναι ότι οι χώρες αυτές προσπαθούν να λάβουν υπόψη τους βέβαια να τους βοηθήσουν ναι, με πλοία κλπ. Μετά έχουμε πολίτες από το νότιο τμήμα της Αφρικής. Μέχρι στιγμής βέβαια δεν έχουμε πολλούς στα σύνορα Λιβύης, την Ισίας Λιβύης, Αιγύπτου. Υπήρχαν όμως στη χώρα, δεν ξέρω πού βρίσκονται. Και οι αρχές του Τσά, της ε, Νιγηρίας, ε, του Μάλι, αναρωτιούνται τι γίνεται, πάνε προς τον Νότο λόγω της βίας που δημιουργείται ακριβώς ε, στις ακτές στο Βορρά ίσως πάνε προς τα νότια. Αλλά μέχρι στιγμής δεν τους έχουμε δει. Και τέλος, επίσης ένα πρόβλημα, γιατί το είδαμε στην Λαπετούσα, ίσως υπάρχουν και πολίτες της ίδια της Λιβύης. Εάν συνεχίσει αυτή η αστάθεια, ίσως χρειαστεί, αισθανθούν την ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν από τη χώρα τους. Όλα αυτά τα εξετάζουμε πολύ προσεκτικά για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά προς το παρόν είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε σαφείς προβλέψεις για το τι θα γίνει ενδεχομένω. Το ξέρουμε και το είπε ο εκπρόσωπος της Frontex, ότι συζητάμε για ένα εκατομμύριο πολίτες από χώρες της Νοτιοαφρικής που μπορεί ίσως να εμφανιστούν, ίσως. Με στιγμής όμως δεν είδαμε τίποτα τέτοιο, δεν πρέπει να παρακολουθούμε τα πράγματα πολύ στενά. Δεύτερο θέμα που μου ερωτήθη, όλα αυτά που σχετίζονται με την νησία. Κύριε παντζέρη, έχετε δίκιο. Η Τινησία ίσως είναι χαρακτηριστικά μια χώρα που θα γίνει μια χώρα επιτυχίας αν δράσουμε σωστά και συνεργαστούμε σωστά με τις τινησιακές αρχές. Έχουμε μιλήσει για το καθεστώς ε, προτιθέμεθα να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι <laughs> για τις διαπραγματεύσεις χρειάζονται δύο. Πρέπει λοιπόν να έχουμε απέναντί μας κάποιες αρχές που να είναι σε θέση να διαπραγματευτούν. Αυτή τη στιγμή οι τυνησιακές αρχές προσπαθούν να βρουν μια λύση συνεργασίες με την αντιπολίτευση που υπάρχει στη χώρα του. Είδαμε ότι ο Πρωθυπουργό παρετήθη. Χθε ορίστηκε ένας άλλος Πρωθυπουργό που ήδη είναι αντικείμενο έντονης κριτικής. Ο Υπουργό ε, Έρευνα και Βιομηχανία επίση παρατηρήθηκε Πρέπει να συνεργαστούμε λοιπόν με τι θρησκευτικέ αρχέ τη ε, προσωρινή κυβέρνηση και θα πρέπει να μα δώσουν μια σαφή εικόνα του πώς μπορούμε από κοινού να προχωρήσουμε. Και μετά υπήρχε ένα τρίτο θέμα. Το τι κάνουμε για να σταματήσουμε την βία. Χημικά όπλα. Το άκουσα από στρατιώτε τα ΜΜΕ, όπω και εσεί έχετε από εκεί τι πληροφορίε σα. Αυτή είναι μια πληροφορία που θα πρέπει να αξιολογηθεί και να επιβεβαιωθεί. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε καμία επιβεβαίωση. Όλοι βρισκόμαστε σε επαφή με τι οργανώσει που μπορούν να το εξετάσουν και ελπίζουμε σύντομα να μάθουμε κάτι παραπάνω σχετικά. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε όμω καμία απόδειξη. Δεύτερον, το γεγονός ότι υπάρχουν 15 μέλη του Συμβουλίου Αυστραλίας που δεν θέλουν να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη γραμμή ε, σημαίνει ότι πρέπει και εμείς να περιμένουμε. Να δούμε πώς θα συνεχιστούν οι συζητήσεις. Αναφερούμε συνεχώς την κατάσταση και πολύ στην συνεργασία όλων των κρατών μελών του Συμβουλίου Ασφαλεία και εδώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πάρα πολύ σημαντική. Ευχαριστώ. Θα σας ευχαριστώ. Η Επίτροπος Μάρσον πρέπει οπωσδήποτε να φύγει. Την ευχαριστούμε λοιπόν για την παρουσίασή τη και τη συμβολή τη και θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Λάτινεν. Παρακαλώ, έστε σύντομος για να έχουμε ένα δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας υπόσχομαι να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Το πρώτο θέμα είναι τι θα γινόταν στην περίπτωση κατά την οποία σας είπα έχουμε έξι σενάρια και έχουμε και ένα έβδομο σενάριο που συνδέει όλα τα έξι πρώτα. Ανάλογα με το σενάριο έχουμε διαφορετικά σχέδια. Ποια θα είναι η αντίδραση του συνοσμού της Frontex. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Το πρώτο, χρειαζόμαστε εκείνο που θα οργανώσει και από την άλλη μεριά τους συμμετέχοντες. Τα κράτη-μέλη δηλαδή θα πρέπει να συμβάλλουν στην ε, ε, εκδήλωση αυτή και θα εμφανίνουμε και τους μεν και τους δε. Είπαμε ότι δεν προσπαθούμε να έχουμε κάποια παλιά σενάρια που να ταιριάζουν για όλους. Έχουμε τόσο πολύ διαφορετικά άτομα όπως ελέγχθη ήδη, τόσο διαφορετικά σενάρια, τόσο διαφορετικά μείγματα μετασταυτικών ροών σε κάθε σενάριο. Δεν υπάρχει μία άγουσα δηλαδή. Και το ίδιο ισχύει για τα λειτουργικά σχέδια. Ο τρόπος λειτουργίας δεν είναι παντού ο ίδιος γιατί εάν υπάρχει ένας τεράστιο αριθμό ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία, δεν πρόκειται να νομίζετε ότι η Frontex θέλει να τους αποκλείσει από το να έχουν την βοήθεια αυτή. Ούτε να σκεφτείτε. Τι γίνεται τώρα. Πότε θα πρέπει να αλλάξει η διαδικασία όταν βρεθούμε στην κρίσιμη κατάσταση. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή. Και αυτή ισχύει και για τη δική μου υπηρεσία. Χρησιμοποιούμε δηλαδή τα μέσα που έχουμε δημιουργήσει. Screening. Αυτό είναι ένα ουσιαστικό τμήμα των δραστηριοτήτων και προσεγγίσεων, όπου ο... η ταυτότητα των ατόμων, ο λόγος για τον οποίο βρίσκεται σε δυσκολίες εξετάζεται εγκάστοτε. Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι Οπωσδήποτε εμπλέκεται και η Πατριαρμοστία Προσφύγων του ΟΕ και εμείς και συντονίζουμε τις δραστηριότητες μας. Θα πρέπει να επαναλάβω ότι δεν αρκούν οι δραστηριότητες στα σύνορα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Δεν είναι αυτή η λύση. Θα είμαστε όμως τμήμα της λύσης, όποια και είναι αυτή. Αναφέρθηκα στους διάφορους τύπους μορροής. Δεν είναι μόνο το θέμα των, ε, της μορφής τους, ε, του ροών, αλλά υπάρχει και αντίστροφη ε, ροή των ατόμων που έχουν ζήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επανέρχονται στις χώρες αυτές. Υπάρχει μια αντίστροφη ροή, όχι σημαντική, αλλά υπάρχει. Καταρχήν, η δυνατότητα δημιουργίας δυναμικού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πώς θα εφαρμοστούν δηλαδή οι δομές αντίδρασης σε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εμπλακεί σε αυτά τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κρίση στα σύνορα. Γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε τρίτες χώρες και να συνεργαστούμε για κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό το ξέρετε γιατί υπάρχει και στον κανονισμό Frontex. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Λάτινεν. Είναι 10 και 20. Όπως λέμε πάντα τίνουμε να ξεπερνάμε τα όρια του χρόνου που διαθέτουμε. Θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια να έχουμε και ένα δεύτερο γύρο. Θα αρχίσουμε το γύρο αυτό. Και προτείνω να μιλήσει ένας εκπρόσωπος από κάθε πολιτική ομάδα και θα συμπεριλάβουμε τους μη εγγεγραμμένους και θα έχουμε ένα δεύτερο γύρο απαντήσεων και βεβαίως οι διερμηνείς θα παραμείνουν λίγο περισσότερο. Μόνο έτσι μπορούμε να το χειριστούμε γιατί διαφορετικά δεν θα τα καταφέρουμε. Σας παρακαλώ, ο κύριος Ιακολίνο έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την παρουσία των εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων για την κατάσταση που είναι ιδιαίτερα επώδυνη στην Βόρειο Αφρική οι κυβερνήσεις προσπαθούν να ανταποκριθούν, ακόμα και οι προσωρινές κυβερνήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να αναλυφθούν ορισμένες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Καταρχήν στο μέτωπο των κυρώσεων έγινε λόγος και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών έγινε λόγος για τον ενεργειακό τομέα και για τις τάχιστες κυρώσεις. Το άσυλο είναι άμεση προτεραιότητα, το κοινό μέτωπο στον τομέα του ασύλου, στη, στον τομέα του Frontex προσπαθούμε να μπορέσουμε να δράσουμε τάχιστα, να δράσουμε με σπουδή. Και βεβαίως η αλληλεγγύη που αναφέρεται στα παχιά μας λόγια, αλλά στην πράξη δεν βλέπουμε αντίκρισμα. Ο κύριος Λάιτινεν θα μεταβεί στη Μάλτα απόψε και ελπίζω να μπορέσει να προβλέψει και τη Λαμπετούζα. Ο κύριος Μπουζούτιλ, διαδικαστικό, από ό,τι κατάλαβα, είπατε θα μιλήσει ένας εκπρόσωπος αναπολιτική ομάδα, αλλά θα ήθελα να τηρήσετε το σύστημα DONT. Και αυτό γίνεται στον πρώτο γύρο, όχι στο δεύτερο. Ναι, αλλά έχουμε θέμα χρόνου. Θα πρέπει να, μιλήσουμε, να μιλήσουν ε, εκπρόσωποι πρόσωποι από τις πολιτικές ομάδες χωρίς να είναι οι 15 που αρχικά προβλέπονταν. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει καλή θέληση έτσι ώστε να έχουμε και γραπτές ε, απαντήσεις από τους ε, εκπροσώπους της ε, Επιτροπής και από τα θεσμικά όργανα. Ο κύριος Ντόρφλερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριος Υπάρχει αυτή η ταινία που λέγεται ότι μας χαιρετά το ζωή συνεχώ. Κοιτάξτε, 16 χρόνια συζητάμε αυτά τα προβλήματα. Δεν άλλαξε τίποτα. Εγώ ήμουν από παλιά βουλευτή και τα ίδια ακούμε. Κύριε Λάιτινεν, αν θέλετε να με ακούσετε σα παρακαλώ, κύριε Λάιτινεν, θέλω να σα πω κάτι. Πριν από πέντε χρόνια, ο κύριο Πουζουτήλη ήταν εδώ, ξεκίνησε στη Frontex. Η Frontex δεν είναι υπεύθυνη για τις ροές των μεταναστών. Αλλά είναι η απόδειξη αυτή το τι κάνει η Frontex. Θέλω να έχω μια απάντηση πώς αντιμετωπίζετε την αξιοπρέπεια των μεταναστών. Λέμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σφαιρικά και διέρετα. Αυτό ισχύει για όλους. Γιατί τη Μάλτα, η Ελλάδα, για τη Λαπεντούζα. Πριν από πέντε χρόνια είχαμε πάει στη Λαπεντούζα και είδαμε πραγματικά ένα φεριχτό το θέαμα που έπαιξε ο Πελουσκόνη μας έδιωξε όλους και έφερε κάποιους επιλεγμένους ε, πρόσφυγες να μας μιλήσουν. Πού είναι η διαφορά ανάμεσα στον Περλουσκόνη και στον κατάφτη. Δηλαδή ο Περλουσκόνη οργανώνει θαυμάσια πάρτι αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ροέ μεταστασίε. αρχίζω και συνεχίζομαι με αυτά που λέγονται εδώ. Δεν αναφέρονται τα προβλήματα. Αποκολύπτονται. Κύριε Μποργέζιο, ο τελευταίος φασιστής ήταν το... Ε, κοιτάξτε. Διακόπτω πρόεδρο τη συζήτηση αυτή μεταξύ των βουλευτών. Η oh. Ιντβελτ, μα δεν μπορώ να δεχτώ αυτές τις προσβολές. Μιλάμε για ένα επώδυνο γεγονός. Δεν έχει νόημα να κάνουμε τέτοιες παρεμβάσεις. Η Συμφωνία Λιβύης Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργήσε πολύ καλά. Μα δεν μπορούμε να, δεν, να κάνουμε τέτοιες παρεμβάσεις. Πρόεδρος, κυρία Ιντβελτ, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι πάρα πολύ αξιοπρεπή όλα αυτά τα πράγματα και έχουμε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε και θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση πριν θέσω τις ερωτήσεις μου. Ε, ως Ευρωπαίοι θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τώρα μπορεί να είμαστε χώρα ε, προορισμού αλλά κάποτε ήμασταν χώρα ε, προορισμού γιατί κάποτε οι άνθρωποι έφευγαν λόγω του πολέμου και έψαχναν μια καλύτερη ζωή αλλού όπου τους υποδέχονταν και δεν τους θεωρούσαν εγκληματίες. Τρεις ερωτήσεις έχω. Πρώτον, ακούω ότι θα εμπλακεί η Europol και θα ήθελα να ξέρω ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος της Europol και πώς συνεργάζεται με τη Frontex. Δεύτερο ερώτημα, ειδικότερα προς τον κύριο Βημό και προς την Ουγγρική Προεδρία. Υπάρχουν και άλλες χώρες, τις οποίες δεν συζητήσαμε σήμερα, όπου βράζουν ε, τα πράγματα. Ε, υπάρχει κάποιος προγραμματισμός, προβλέπουμε κάπως ε, τη συνδρομή μας προς ε, τέτοιου είδους χώρες ή περιμένουμε πρόσφυγες από τις χώρες αυτές. Και μία τελευταία ερώτηση. Κρίμα που η Επίτροπος έφυγε. Ανέφερε ενδεχομένως οι υπόλοιποι ομιλητές να, να μπορούν να απαντήσουν οι υπόλοιποι. Ανέφερε 25 εκατομμύρια ευρώ ως ε, ταμείο κατεπήγων. Μου φαίνεται πάρα πολύ λίγο για μια κατάσταση τέτοιας κλίμακας. Ίσως οι υπόλοιποι να μπορούν να πούν κάτι σε σχέση με το πώς διατίθενται τα χρήματα αυτά και τι άλλους πόρους μπορούμε να αναζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κέλλερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ένα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ξέρω τώρα ποιος μπορεί να το απαντήσει. Υπάρχουν πρόσφυγες στη Λιβύη, τους οποίους εμείς στείλαμε πίσω από την Ιταλία και αναρωτιέμαι τι προστασία δίνουμε στους ανθρώπους αυτούς. Δεν αισθανόμαστε υπεύθυνοι για τους ανθρώπους αυτούς που τους στείλαμε πίσω στη Λιβύη. Ερώτημα προς τη Frontex. Είπατε ότι δεν εμποδίζεται τον κόσμο να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να μου πείτε ακριβώς τι κάνει η Frontex τελευταίες εβδομάδες στη Μεσόγειο εφόσον ε, τώρα πια μπορεί να μην έρχονται μετανάστες, αλλά τι νομίζετε ότι θα γίνει ε, ή τι έγινε στο παρελθόν όταν έρχονταν οι άνθρωποι αυτοί. Και επίσης, ε, όταν θα, θα τελειώσει η διαδικασία συναπόφασης, τέλος πάντων πότε θα τελειώσει, γιατί τότε μπορούμε να περάσουμε στην κατεπίγουσα διαδικασία. Και μια, ένα ακόμη ερώτημα έχω να θέσω, μια και συζητάμε τις εξελίξεις ε, στην Ανατολική Ευρώπη. Ε, βλέπατε τότε τα πράγματα ως απλώς μεταναστευτική ροή ή βλέπατε επίσης και τη θετική ε, πλευρά των όλων, του, του όλου πράγματος. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης για ένα λεπτό. Βρέσει λιγότερο από ένα λεπτό, δύο μικρές ερωτήσεις Έχω παρακολουθήσει τις δηλώσεις που έχουν γίνει από την κυρία Νάστον και από πολλούς άλλους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε, νομίζω, σε μια γλώσσα μη κατανοητή από τους πολίτες. Θέλω έτσι στο πρακτικό επίπεδο να ρωτήσω ποιες χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να δεχθούν μετανάστες οι οποίοι ενδεχομένως να έρθουν σε μεγάλους αριθμούς από αυτές τις αραβικές ε, χώρες και να τους δεχθούν κατά τρόπον που να τους ενσωματώσουν στις κοινωνίες τους, όχι σαν ένα περιστατικό αντιμετώπισης μιας πολεμικής κατάστασης. Και δεύτερη μου ερώτηση είναι για το resettlement co-decision, is this on the agenda? Thank you very much. Thank you. Mrs. Mobile for the non Η κυρία Μορβάη για τους μη Ένα λεπτό. Δύο σύντομες ερωτήσεις έχω προς την Ουγγρική Προεδρία και σε όποιον άλλον θέλει να την απαντήσει. Γιατί είναι τόσο φυσικό ε, οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι, ε, οι, νοσο, οι νοσοκόμοι, οι μικροί επιχειρηματίες που πρέπει να πληρώσουν ε, το τίμημα των ε, δικτοταριών που καταραίουν. Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο είδους οικονομικός διακανονισμός ώστε τα τα παγωμένα αυτά ε, ποσά που οι δικτάτορες κλέψανε από τους λαούς τους θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν το κόστος ε, όλων ε, αυτών των τον άσυλο και των προσφύγων. Η κυρία Μάλμστρομ είπε ότι οι φυσιολογικές συνθήκες θα αποστέλλονταν οι άνθρωποι δεν θα αποστέλλονταν ποτέ πίσω ε, στις ε, χώρες τους. Όμως ε, μιλάμε για δημοκρατική μετάβαση. Εφόσον θα γίνουν δημοκρατίες, ελπίζουμε σύντομα οι χώρες αυτές, για ποιο λόγο να μην μπορούν να επιστρέψουν στις δημοκρατικές τους χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, Μάλιστα. Τώρα, Deon System για τις μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες, για το ΕΛΚ, ο κύριος Παπα-Νικολάου θέλει να πάρει το λόγο. Σύντομες ερωτήσει κύριε Πρόεδρε και σα ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Κύριε Λάιτινεν, είπατε ότι η κατάσταση αυτή συνδέεται με τα προβλήματα που έχουμε για τις ζωές και στην Ελλάδα και στα κρατημέλη. Η Ελλάδα πριν από δύο μέρες, η Τουρκία συγγνώμη, πριν από δύο μέρες πριν ανήγγελε ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα εφαρμόσουν τη νέα συμφωνία που προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε, όπως είπε και η Κομισιόν, ε, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις επειδή δεν τους δίνουν απελευθέρωση από θεώρηση διαβατηρίων. Ρωτώ λοιπόν, υπάρχει μια ευρωπαϊκή αντίδραση για τη δήλωση αυτή της τουρκικής πλευράς. Σας ευχαριστώ κύριος Λαμπρινίδης. Ένα λεπτό. Πολύ σύντομα πρόεδρε. Η κατάσταση κρίσης, σαν αυτή που έχουμε, καταδεικνύει με τον τρόπο αυτό που ζητάνε εδώ και πολύ καιρό. Δηλαδή τα προβλήματα και τα όρια τους δεύτερους Συμφωνίας ε, Δουβλίνου. Ε, καταλαβαίνω ότι ορισμένα κράτη-μέλη και ε, στο Συμβούλιο δεν ε, θέλουν να διευρυνθεί η εγγύηση αυτή για την επανεγκατάσταση. Αυτό που κάνουμε είναι ότι στέλνουμε το μπαλάκι πέσει σε εκείνους που είναι επιτόπου στα σύνορα, οι οποίοι μας το ξαναστέλνουν εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Λοιπόν. Ε, κύριε Μάρσο, δεν να απαντήσει, αλλά εγώ ρωτάω τώρα. Στο Συμβούλιο ορισμένοι δέχτηκαν να υποδεχθούν ζητούντες άσυλο όταν φτάσουν στα σύνορά τους. Θεωρώ όμως ότι το να δώσουμε ε, βοήθεια οικονομική σε εκείνους που είναι στα σύνορα δεν θα βοηθήσει την Μάλτα, την Ελλάδα, την Ιταλία να αντιμετωπίσουν αυτές τις τεράστιες μεταστατικές ροές. Όσον αφορά λοιπόν πραγματική αλληλεγγύη δεν θα πρέπει να ξυπνήσει το Συμβούλιο και να τελειώσει μια κατάσταση που είναι καταστροφική και για τα καρατημένη και για εκείνους που ζητούν άσυλο. Ευχαριστώ, ο κύριος Μοζινιόρ. Ευχαριστώ. Διαπιστώσαμε ότι η πολιτική μας, η προτιμησιακή μας πολιτική υπέρ των δυνατών ανδρών απέτυχε ικτρά. Τι θα κάνει το Συμβούλιο έτσι ώστε να έχουμε ισχυρούς θεσμούς αλλά όχι ισχυρούς άνδρες. Μιλήσαμε για την Ένωση για τη Μεσόγειο, τη διαδικασία της Βαρκελόνης, τη Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών και ούτω καθεξής τι σχέδια έχουν Επιτροπή και Συμβούλιο έτσι ώστε να υπάρξει μια κοινωνικο-οικονομική ανάκαμψη της Μεσογείου. Επίσης ε, διαπιστώνουμε ότι οι υπηρεσίες της Ένωσης δεν μπορούν να προβλέψουν τα τεκτενόμενα και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια στις προβλέψεις. Εγώ δεν δέχομαι τα συγχαρητήρια για το τι έγινε. Εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα. Η κυρία Ρομέρο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ξέρει τι συμβαίνει. Γιατί οι επαναστάσεις που ζούμε στη νότια όχθη της Μεσογείου είναι η δική μας επανάσταση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τίποτα πια δεν θα είναι το ίδιο. Δεν πρόκειται για θέμα επικοινωνίας. Είναι εσχρό το ότι γνωρίζουμε τι συμβαίνει και μιλάμε μόνο για τα προβλήματα ενέργειας ή για τα προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι έσχος αυτό δεν είναι θέμα επικοινωνίας, είναι θέμα πολιτικής οπτικής. Εγώ λυπάμαι που είμαι Ευρωπαία πολίτης. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να κάνει πολύ ε, περισσότερα. Το Frontex θα πρέπει να αλλάξει, να αλλάξει όνομα διότι μιλάμε για ε, μια δημοκρατική διαδικασία. Οι κυβερνήσεις αυτές οδεύουν προς τη δημοκρατία και εάν εμείς δεν μπορέσουμε να έχουμε μακρύ ορίζοντα δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Αλφάνο, για ένα λεπτό, τελευταίος γύρος. Ευχαριστώ δεν πρόκειται για, ε, για μία ε, φάρσα. Μιλάμε για την αλήκη στη χώρα των θαυμάτων. Λέμε τι συνέβη στη Λιβύη. Μα τι κάναμε εμείς στην ουσία, υποστηρίξαμε αυτές τις κυβερνήσεις μέσα στα πλαίσια ε, των προτιμησιακών σχέσεων και των εμπορικών σχέσεων. Όταν μεταβήκαμε στη Λιβύη, τι κάναμε. Μιλήσαμε για μία διαδικασία συναλλαγών σαν να ήμασταν τουρίστες και τίποτα άλλο. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο υπαριθμόν δύο της κυβέρνησης της Λιβύης μας έστελνε από το εν μεν στο δε μέρος χωρίς όμως να καταφέρουμε τίποτα. Είναι μία αποτυχημένη πολιτική. Δεν ε, σας διέκοψα, μη με διακόπτετε. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ψηφοφόροι μας μας λένε ότι στην ουσία βάλαμε πρώτα τις εμπορικές συμφωνίες πριν από τη ζωή εκατομμυρίων πολιτών. Και αυτό το κάναμε και στην Κίνα, το κάνουμε και στη Λιβύη. Αυτή τη στιγμή σκοτώνονται αυτοί οι άνθρωποι από τον Καντάφη. Λυπάμαι οι Ιταλοί συμπατριώτες μου θα πρέπει να δεχτείτε αυτές τις επικρίσεις διότι όταν ο, Κεντάφ, ο Καντάφη σκότωνε του συμπολίτες του, ο Μπερλουσκόνη είχε πει «Ας μην ενοχλούμε τον ε, Καντάφη». Αυτό είχε πει τότε ο Μπερλουσκόνη. Υπάρχουν ε, και άλλα μέλη που θα ήθελαν να λάβουν το λόγο, θα πρέπει όμως να κατανοήσετε ότι δεν μπορούμε να υπερβούμε κατά πολύ το χρόνο μας, αν θέλουμε απαντήσεις ε, από τους προσκεκλημένους μας. Γι' αυτό θα πρότεινα το εξής. Όσοι δεν λάβατε το λόγο να υποβάλλετε τις ερωτήσεις γραπτός, έτσι ώστε να έχουμε γραπτές απαντήσεις και από την εξωτερική υπηρεσία και από την Κομισιόν. Τώρα θα έχουμε τον τελευταίο γύρο από τον πρέσβη Γιώργος, μετά τον Γενικό Γραμματέα και τον κύριο Λάτινεν. Ο κύριος Γιώργος έχει το λόγο. Σας παρακαλώ κύριε Ταβάρες είναι ιστορική ε, σημασία αυτό, γιατί οι Ούγγροι ε, φορολογούμενοι πρέπει να πληρώσουν για αυτά. Θέλω να σε υπενθυμίσω ότι η πρώτη μεγάλη ε, δραστηριότητα προ, προστασία των προσφύγων σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν το 56 για τους Ούγγρους πρόσφυγες. Μα αυτό δεν ήταν διαδικαστικό, λέει ο πρόεδρο, ήταν θέμα της συζήτηση. Α στηρίξετε την διαδικασία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και ο Γιώργος. Για το τελευταίο θέμα, δεν θέλω να σχολιάσω τις απώλειες χιλιάδων ζώων στην Ουγγαρία το 1956. Απλώς δεν θέλω να σας αναφέρω κάποια συγκεκριμένα θέματα. Κατά πόσο πόσον προχωρήσει η διαδικασία συναπόφασης, τι να σας πω, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά θα πρέπει να συνεργαστούμε νομίζω με το Κοινοβούλιο για την, ε, το θέμα της επανεγκατάστασης. Ε, η Ουγγρική Προεδρία προσπαθεί να επιταχύνει την κατάσταση. Κατά πόσον μπορούν να υπάρξουν επίγουσε καταστάσει και σε άλλες χώρες, δεν τολμώ να προβλέψω τίποτα. Κατά πόσον οι διαδικασίες στον αραβικό κόσμο θα προχωρήσουν, δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά η Ευρώπη πρέπει να μπορεί και από ό,τι ξέρω μπορούσε μέχρι στιγμής να αντιδράσει για να μπορέσει να βοηθήσει τις δημοκρατικές διαδικασίες. Είναι απόλυτα σαφές ότι αφενός πρέπει να εξασφαλίσουμε την τροφοδότηση με ενέργεια, την εσωτερική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ταυτόχρονα να βοηθήσουμε τις δημοκρατικές δυνάμεις που προωθούν αυτές τις εξελίξεις στις εν χώρε και θα πρέπει με το δικό μας δημοκρατικό παρελθόν να φροντίσουμε οι χώρες αυτές να έχουν δημοκρατικό μέλλον και η οικονομική και κοινωνική κατάσταση που δεν θα προωθούν εκατομμύρια ανθρώπων στο να προσπαθούν να μεταβούν στην Ευρώπη. Τώρα, όσον αφορά τον, το πάγωμα των περιουσιών, αυτό ε, εφαρμόζεται ήδη εχθές ε, ληφθεί απόφαση. Διεθνή συμφωνία θα έχω να σα πω ότι το Συμβούλιο γενικά ενέκρινε τα αποτελέσματα διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Τουρκία, και τώρα τα δύο μέρη θα πρέπει να ε, υπογράψουν και να επικυρώσουν τις εν συμφωνίες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο για οποιασδήποτε δηλώσει έγιναν, θα πρέπει να δούμε τις εξελίξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια ενδιαφέρεται πάρα πολύ για αυτή την συμφωνία επανεγκατάσταση και δίνει το, Κομισιόν, το Συμβούλιο συγγνώμη, στην Κομισιόν ε, το πράσινο φως κατά κάποιο τρόπο για να περάσει σε διάλογο. Αλλά δεν προβλέπεται τίποτα αυτή τη στιγμή για απελευθέρωση από την υποχρέωση θεώρησης. Αλληλεγγύη. <clears throat> Ανέφερα ότι η κατάσταση είναι πολύ πολύπλοκη συζητήσει το Συμβούλιο αναγνώριζα πλήρω την πρόκληση που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την Μάλτα και την Ιταλία και ορισμένε χώρε μέλη χρειαζόνται σαφεί αναφορές όσον αφορά τι δικέ του δραστηριότητε για νόμους και παράνομε μετανάστες και είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια δίκαια και οριζόντια εικόνα. Κατανομή του βάρου υπάρχει στην πράξη Κανένας δεν έχει πει όχι. Ένα παράδειγμα, η Σουηδία το 2010 υπεδέχθη πάνω από 40.000 μετανάστες πρόσφυγες από το Ιράκ και 5.000 ε, πρόσφυγες από τη Σερβία χωρίς να ζητήσει καμία ελεγγύη. Θα πρέπει λοιπόν να βάλουμε υπόψη μας όλες τις προσπάθειες κρατών μελών και συζητάμε την κατάσταση και τα προβλήματα γενικά από την ελληνική. Και όσον αφορά όλα τα στοιχεία των σχέσεων με τις γειτονικές χώρες, ε, φαντάζομαι ότι ο Γενικός Γραμματέας θα αναφερθεί στα θέματα αυτά, κατά πόσον η διαδικασία της ευρωπαϊκής ε, πολιτικής ε, γειτνίασης υπάρχει αυτή η στιγμή όπως είπατε, συζητιέται. Ευχαριστώ, κύριος Δημό, έχετε λόγο. Mm. Once θα είμαι και πάλι πάρα πολύ σύντομο, Συνεχίζοντας αυτά που είπε η Ουγγρική Προεδρία, όπω γνωρίζετε, είναι διτή η προσέγγιση μας. Πρώτον, προσπαθούμε <clears throat> να υπάρξει ένα πακέτο μέτρων ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και είπα τι εκπρόσωπος ε, να καταλήξουν ε, ε, στις 24 με 25 Μαρτίου για το πακέτο αυτό. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας εξακολουθεί να υφίσταται θα γίνει μια αναθεώρηση βέβαια τον Απρίλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας πει τις τελευταίες της ιδέες για το θέμα αυτό. Αυτές οι δύο διαδικασίες βέβαια αλληλεπιδρούν. Και όπως δικαίως υπόθηκε, πρόκειται για ένα φαινόμενο τόσο μεγάλης εμβέλειας σε σχέση με αυτή την προσπάθεια εκδημοκρατισμού χωρών που δεν είχαν δημοκρατία για μεγάλο χρονικό διάστημα, που πρέπει ε, λίγο να δούμε τι μέτρα μπορούμε να λάβουμε προκειμένου να βοηθήσουμε τις χώρες στον εκδημοκρατισμό. Αυτό δεν είναι μόνο βραχυπρόθεσμα τα μέτρα αυτά. Πρόκειται για ισχυρά μακροπρόθεσμα μέτρα που θα δώσουν τη δυνατότητα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξη των χωρών αυτών. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι μόνη τη την περασμένη Τετάρτη είχαμε μία συνάντηση της ε, των, ε, του ΟΗΕ, ε, των διαφόρων οργανισμών του ΟΗΕ σε επίπεδο διεθνούς κοινότητας γίνονται πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες κινητοποίησης. Επίσης ε, είχαμε επαφές και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης που ότι θα άλλαζε μέχρι και το καταστατικό της για να μπορέσει να βοηθήσει. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει τεράστια κινητοποίηση πολλών και διαφορετικών εταίρων προκειμένου να βοηθηθεί η κατάσταση. Βέβαια θα χρειαστεί χρόνος και πρέπει να δούμε και τις εξελίξεις επιτόπου. Με ρωτήσατε τι κάνουμε από άλλες χώρες. Βεβαίως ε, παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ ε, προσεκτικά, όμως πρέπει να γνωρίζουμε και το έχουμε πει πολλές φορές ότι κάθε χώρα ε, ακολουθεί μια διαφορετική διαδικασία όσο εξελίσσονται ε, τα πράγματα. Η Τινήσια και η Αίγυπτος ακόμη ε, διέρχονται ε, πολιτική μεταρρύθμιση. Υπάρχουν επίσης στο Ομάν, στο Κατάρ, στην Ιεμένη πολλές εξελίξεις, τις οποίες παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και βέβαια θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα αν χρειαστεί. Αυτό θα είναι τεράστια σημασία ε, και μεγάλη προτεραιότητα τη ε, ημερήσια διάταξη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Με ρωτήσατε για το θέμα της διαδικασίας ασύλου. Στην περίπτωση της μετανά... των μεταναστών της Λαμπεντούσα, βεβαίως ισχύει η διαδικασία του ασύλου. Μιλάμε τώρα προσπαθούμε να δούμε, για το πώς, να δούμε πώς αλλάζει η πολιτική κατάσταση της χώρας από την οποία προέρχονται, προκειμένου την Τινησία. Πρέπει λοιπόν αναλόγως να προσαρμόσουμε και τη διαδικασία ασύλου υπό το φως των εξελίξεων στη χώρα αυτή. Και πρέπει να δούμε τι θα κάνουν και τα κράτη-μέλη όσο προχωρεί η διαδικασία. Και τε, ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τέλος, από τη Frontex, ο κύριος Ιλκα Λάτινεν. Κυρία Γκόμες, είναι διαδικαστικό. Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να πω ότι είναι εξωφρενικό το γεγονός ότι ε, η συνάδελφος έκανε την ε, δήλωση αυτή της αποστολής ε, που πήγε στη Λιβύη έφυγε στο τέλος της πρώτης μέρας. Δεν ήταν εκεί στις επισκέψεις που κάναμε στα κέντρα κρατήσεων και είναι πραγματικά εξωφρενικό το γεγονός ότι έκανε τα σχόλια που έκανε. τα στοιχεία που συλλέξαμε στην επίσκεψη αυτή μας έδωσε τη δυνατότητα, τη δυνατότητα να, ε, να εκπονήσουμε την ε, σύσταση που εκπονήσαμε πέρσι ε, τον Ιανουάριο. Είναι απαράδεκτη η δήλωσή της. Πρόεδρος. Σύντομα θα κάνουμε μια συζήτηση, ε, κυρία Γκόμε, για το τι ακριβώ είναι διαδικαστικό αίτημα. Πρέπει να το συζητήσουμε. Τι είναι διαδικαστικό αίτημα σύμφωνα με το εσωτερικό κανονισμό δεν είναι να ξαναρχίζουμε τη συζήτηση, δεν είναι να κάνουμε μια δήλωση, δεν είναι να αντιλέγουμε σε οποιονδήποτε συνάδελφο. Είναι απλώς να ε, δούμε κατά πόσο έγινε σεβαστός ένας κανόνας του εσωτερικού κανονισμού του Κοινοβουλίου και αν δεν ελήφθη σωστά υπόψη. Οπότε λοιπόν ας ακούσουμε την τελική τοποθέτηση ε, του Διευθυντή της Frontex, του κυρίου Λάιτινεν. Δεν, βρίσκω σωστό. Εσείς είπατε ότι έκανε λάθος η συνάδελφη. Εφόσον έκανε λάθος εκείνη, τότε ας απαντήσω κι εγώ στο λάθο της συναδέλφου. Πρέπει να απαντήσω. Πρέπει να απαντήσω. Ε, αν τα πράγματα είχαν όπως έπρεπε να έχουν, θα είχα παραμείνει και την ε, τελευταία ημέρα. You got the floor. Κύριε Λατίνεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Έχω λοιπόν τον τελευταίο λόγο και πρέπει να είμαι περήφανος γι' αυτό. Τρία σημεία θα ήθελα να επισημάνω. Πρώτον, το θέμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ε, με όλα τα μέσα που έχουμε στις επιχειρήσεις μας, ε, υπό την ηγεσία και τον έλεγχο των κρατών μελών και υπό τον συντονισμό της Frontex. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να πω. Το δεύτερο που ήθελα να πω αφορά ε, την περίπτωση της Λαμπεντούζα, την ε, παράνομη μετανάστευση από την αρχή του χρόνου από την Τινησία, ειδικότερα κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες προς τη Λαμπεντούζα. Ε, αναφέρθηκε από την, από την κυρία Κουτέρες την, την περασμένη εβδομάδα και από την Επίτροπο Μάλμστρομ Πρόκειται για άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Αυτό αναφέρθηκε ευθαρσώς. Υπήρξαν ελάχιστες περιπτώσεις μεταξύ των 6.000 που υπήρχε αμφιβολία για τη χορήγηση ασύλου. Είναι οικονομική παράνομη μετανάστες αυτή την περίπτωση. Είναι λοιπόν διαφορετικά τα μόντιο περάντι όπως ως προς το θέμα αυτό. συμμετείχαμε με αεροπορικά μέσα στην περιπολία των ε, χωρικών υδάτων της Ιταλίας, ενισχύοντας την Ιταλική ικανότητα ε, στην περίπτωση αυτή και αποστήλαμε πυρογνώμονες για να βοηθήσουμε τους εμπειρογνώμονες, τους Ιταλούς ε, στο screening και στην παρακολούθηση. Και το ίδιο κάνουμε όσον αφορά τις ε, ε, διαδικασίες επαναπατρισμού, οι οποίες εξακολουθούν να συμβαίνουν μεταξύ Ιταλίας και την ε, Τελευταίο σημείο για την Europol. Δεδομένου ότι υπήρχε ένα διοικητικό κενό στην Τινησία που οδήγησε σε αυτή την κατάσταση, εγώ συμφώνησα ότι χρειάζεται η βοήθεια της Europol. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε. Ουσιαστικά με την κινητή τους ε, ομάδα ε, χρησιμοποιούν τις, προ... τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους γιατί εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε τα στοιχεία αυτά σε αυτή τη φάση. Αυτά ήταν τα τρία σημεία που θα ήθελα να θέσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών που με προσκάλεσε γιατί είναι πραγματικά μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για να μοιραστώ τις σκέψεις μου μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς ε, εσάς για όλες τις προσπάθειες που κάνατε. Ευχαριστώ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ τους βουλευτές για την κατανόησή τους για τους χρονικούς περιορισμούς που έθεσα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους τους διεμηνείς ε, για τα επιπλέον 20 ε, λεπτά που λάβαμε για την έκτακτη αυτή συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστώ πολύ και καλή σας μέρα.